να δράσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζει τις μονομένες κυρώσεις αμέσως για να πιέσει πιο άμεσα το καθεστώς. Ακόμη και έτσι πιστεύω ότι δεν θα ήταν έξυπνο να κόψουμε κάθε επαφή με την κυβέρνηση Νικαράγουα, οι εκλογέ, εκλογές, εκλογική μεταρρύθμιση και το τέλος της καταστολής θα έλθουν μόνο μέσω του διαλόγου και για ε, να αρχίσει εκ νέου διάλογος η Ευρωπαϊκή Διπλωματία μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ας πιέσουμε το καθεστώς αλλά ας μην κλείσουμε τις πόρτες. Ας είμαστε ευφυείς και ας δράσουμε με χρήσιμο τρόπο. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Λόπες Αγγιλά. Ευχαριστώ κύριε Υπατεκπρόσωπε όπως και στην περίπτωση της ε, Βενεζουέλας, όλες ε, τις ε, καταγγελίες τις ενστερνίζομαι που αφορούν τα βασανιστήρια, τις εξοδικαστικές εκτελέσεις στην Καράγουα κτλ. Όμως υπάρχει μια διαφοροποίηση από τη Βενεζουέλα. Εδώ και πολύ καιρό μετά από τη Σαντινιστική Επανάσταση ο πρόεδρος Ορτέγα βγήκε με εκλογές και επομένως σε κάθε εκλογές στην Καράγουα είχαμε εκλογική αποστολή του του Κοινοβουλίου. Η τελευταία έκθεση ήταν ιδιαίτερα επικριτική. Εσεί αναφέρετε δυνατότητα ότι στο μέλλον ε, θα μπορούσαμε να έχουμε εκ νέου ελεύθερε διαφανεί ε, και πραγματικά δημοκρατικέ εκλογέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στείλει μια εκλογική αποστολή για να το εγγυηθεί, αλλά πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά. Θα πρέπει να ασκήσει όλο το διπλωματικό τη βάρο η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να έχουμε το συντομότερο μια αξιόπιστη εκλογική διαδικασία στην Βενεζουέλα για να επιστρέψει η δημοκρατία και και ε, να δούμε και τον πρόεδρο Ορτέγα να εκλέγεται, ε, εάν προκύψει αυτό, μέσω δημοκρατικών εκλογών. Mr. Wallace, one minute. Wallace, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, η επιλεκτική ακοή ε, είναι κάτι το προβληματικό. Κατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων έχουν ε, συγκεντρωθεί στη Μανάγουα για να ε, εορτάσουν το καθεστώς του Σαμόζα το 79, την ανατροπή του καθεστώτος Σαμόζα το 79. Έχουμε λοιπόν μια εκλεγμένη κυβέρνηση αλλά υπήρξαν διαμαρτυρίες από ακροδεξιούς η CIA και αυτή αναμίχθηκε. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, χρηματοδότησαν ΜΚΟ και άλλαξαν τα στοιχεία κατά της κυβέρνησης. Ε, κάποιες ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έγιναν όπλα για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Κοιτάξτε, αυτή η χώρα, όπως και πολλές χώρες της Νότιας Αμερικής, έχουν υποφέρει πάρα πολύ για πολλά χρόνια. Η ανάμειξη των ε, Ηνωμένων Πολιτείων οδήγησε τους ανθρώπους να πάνε στα σύνορα με το Μεξικό η ε, χώρα έχει καλυφθεί από εταιρείε των ΗΠΑ και δεν υπάρχει καμία δικαιοσύνη. Κύριε Μπορέλ, έχει έρθει η στιγμή η Ευρώπη να υψώσει τη φωνή της και να επιτρέψει στους πολίτες της Νικαράγουα, της Βενεζουέλας και άλλων ε, κρατών στην περιοχή να αποφασίσουν μόνοι τους για το μέλλον τους. Ο κύριος Καστάλντο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου να εκφράσω την υποστήριξή μου προς τον λαό της ε, Νικαράγουας ε, που έχει ζήσει μια τραγική κρίση ανθρωπιστική, οικονομική, ε, πάρα πολύ τραυματισμένη. Όλοι αυτοί οι διαδηλωτέ είναι η τραγική κρίση που μένεται εδώ και αρκετό καιρό στην Νικαράγουα. Έχει ακολουθηθεί μια βίαιη στρατηγική έναντι των ειρηνικών διαδηλετών. Αυτό ε, το έχουν αποφασίσει κυβερνητικά στελέχη. Είναι ε, ένα πλήγμα παρά κατά της ε, δημοκρατίας και της ελεύθερης ε, ζωής. Οι παραβίαση των δικαιωμάτων και η κατάχρηση της εξουσίας από πλευράς ε, του Ορτέγκα, του οικογενειακού του καθεστώτος παραβιάζουν την δημοκρατική τάξη της χώρας. Οι φυλακισμένοι ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες και γι' αυτό καλούμε τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να εγγυώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τους συναδέλφους να εφαρμόσουν Μόνο αν υπάρχει σεβασμός ε, των συμφωνιών, μόνο έτσι θα υπάρξει μία διέξοδος από την τραγική αυτή κρίση και κύριε είπατε εκπρόσωπε, εμείς αυτό θα το στηρίξουμε. Και για να... Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η διαδικασία Catch the Eye και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους σας. Ένας, μια δημοκρατική αντιμετώπιση της κρίσης απαιτεί εκλογές, εκλογικές και μεταρρυθμίσεις για να μπορούν οι πολίτες να αποφασίσουν για τη μοίρα τους. Και νομίζω επ' αυτού ε, συμφωνούν όλοι. Αλλά δεν πιστεύω ότι γι' αυτό φταίνε η CIA ή οι εταιρείε της μπανάνας. Αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση καταστολής, παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευράς του καθεστώτος Ορτέγκα. Και το γεγονός ότι ο Ορτέγκα παλιά, αλλά πραγματικά πολύ παλιά, ήταν αντάρτης, γκοριλιέρο και αγωνιζόταν για την ελευθερία της χώρα ε, αυτό δεν αλλάζει τίποτα στην τρέχουσα κατάσταση. Όλοι σας λοιπόν θέλουν το καλύτερο για τους πολίτες της Νικαράγουα, πόσο μάλλον εγώ. Αλλά η πολιτική δεν είναι το να εκφράζουμε ευχές και επιθυμίες. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Και μερικοί είπαν ε, να αρθεί η εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με την Ικαράγουα. Νομίζω η ε, αναστολή αυτής της συμφωνίας θα δημιουργούσε περαιτέρω πόνο και δυσκολίες για τους πολίτες της Νικαράγουας και όχι μόνο στην χώρα αυτή αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό είναι καλή ιδέα. Τότε γιατί να μην ανασταλεί η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την έχουμε αναστείλει ε, για να μην ε, υποφέρουν οι πολίτες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι η βοήθεια που δίδεται είναι να μην, ε, από αυτή να μην υποφελείται το καθεστώς, αλλά να στηρίζονται οι πρόσφυγες, παραδείγματος χάρη, στην Κωνσταντίνα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γιατί δεν ανέστηλε τις δραστηριότητές της για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Παραμένουμε πιστοί και τηρούμε τις ε, ε, υποχρώσεις μας, συμβατικές υποχρώσεις μας. Βεβαίως και θέλουμε ε, πρόορες εκλογές κατά τα μέσα του 18 κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων η αντιπολιτεύση επέμεινε σε πρόορες εκλογές ένα αίτημα το οποίο βία απέρριψε ο Ορτέγκα. Δεν έχουν υιοθετηθεί εκλογικές μεταρρυθμίσεις και αν δεν γίνει αυτό, τότε η εκλογική διαδικασία δεν θα βοηθήσει καθόλου. Η δική μας η προτεραιότητα πρέπει να είναι η εφαρμογή εκλογικών μεταρρυθμίσεων με βάση τις συστάσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην τελευταία αποστολή ε, παρακολούθησης της κατάστασης. Γιατί δεν έχουμε επιβάλει κυρώσεις κατά το Ορτέγκα. Κοιτάξτε, οι Ηνωμένε Πολιτείε και ο Καναδάς έχουν επιβάλει ε, συγκεκριμένες ατομικές κυρώσεις ε, κατά του Ορτέγκα και της οικογένειάς του. Εμείς ακόμα δεν το έχουμε κάνει αυτό. Είναι κάτι που θα πρέπει να το σκεφτούν τα κράτη-μέλη και δεν το αποκλείω να συμβεί στο μέλλον. Όμως, οι κυρώσεις, ε, κατά κύριο λόγο, ε, έχουν στόχο να προκαλέσουν κάποια αλλαγή και γι' αυτό πρέπει να τα σταθμίσουμε τα πράγματα. Θα στείλουμε ε, Επιτροπή Παρακολούθηση των Εκλογών στην Νικαράγουα. Όσο έχει τώρα η κατάσταση, λόγω της πίεσης που ασχολείται τη βία και επειδή δεν υπάρχει κράτο δικαίου δεν έχει νόημα να στείλουμε τέτοια αποστολή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ασκήσουμε πολιτική και διπλωματική πίεση για να απελευθερωθούν οι κρατούμενοι, όχι όλοι βέβαια, αναφέρθηκε ενδεικτικά ένα ή δύο, υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι και πρέπει να σας ενημερώσω ότι ο επικεφαλής αντιπροσωπείας μας στην Ικαράγουα έχει επισκεφθεί οικογένειες ε, αυτών των ε, φυλακισμένων που αναφέρθηκαν τα όνοματά τους, έχουν επισκεφθεί τους γονείς τους. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να ασκούμε πίεση γιατί πιστεύω ότι στην περίπτωση της Νικαράγουας έχουμε συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι' αυτό. Και αυτό είναι σαφέστατα ένα θέμα που αφορά ένα καθεστώς το οποίο δεν περνάει ε, καμία ε, δοκιμή για το πόσο σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αγαπητοί βουλευτές, Ε, εκφράστηκε η επιθυμία να προσθεθούν ονόματα στον κατάλογο των ανθρώπων κατά των οποίων επιβάλλονται ατομικές κυρώσεις. Επ' αυτού όμως πρέπει να συμφωνήσουν ομόφωνα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εμείς θέλουμε την υποστήριξή σας για να αντιμετωπίσουμε ε, στην Ικαράγουα μία κατάσταση που το είπα και πριν είναι τόσο κακή όσο και στη Βενεζουέλα. Αλλά όμως δεν μιλάμε τόσο για την Ικαράγουα. Να, σήμερα όμως το κάναμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε. Έχω λάβει τέσσερις προτάσεις ψηφίσματος κατόπιν αυτή τη συζήτησης από τους Σοσιαλιστές Δημοκράτες, Επρασίνους, ΕΛΚ, ΡΙΝΙΟΥ και Ευρωπαίοι Στρατηγικοί Μεταρρυθμιστέ. Φτάνουμε στο τέλο τη συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Το Επόμενο σημείο της μέσης διάταξης είναι η δήλωση ε, του του εκπροσώπου της ε, Επιτροπής και Προέδρου της Επιτροπής και ύποτου εκπροσώπου ε, σε ό,τι αφορά τις, τη βία καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στα Ιράν. Σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να ζητήσετε Catch the Eye και τη διοίκηση της γαλάζιας κάρτας μέσω των συνήθων διόδων εγγραφής. Μπορείτε να βρείτε οδηγίες στην είσοδο της αίθουσα Ολομέλειας και επιθυμίζω ότι οι ερωτήσεις μέσω γαλάζιας κάρτας επιτρέπονται μόνο μετά τις ε, ομιλίες των πολιτικών ομάδων. Το λόγο έχει ο κύριος Μπορέλ, το εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εξότιμα μέλη. Γνωρίζετε όλοι ότι το Ιράν βρίσκεται εν μέσω μιας εξαιρετικά σοβαρής οικονομικής κρίσης με ελλείψεις ε, βασικών αγαθών, φαρμάκων, έχουμε ψηλά επίπεδα πληθωρισμού, ανεργίας και όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε διαδηλώσεις. Εγώ και η υπηρεσία μου έχουμε παρακολουθήσει τις εξελίξεις ε, εκ του σύνεγγυς από τις 15 Νοεμβρίου προσπαθούμε να αποκτήσουμε αξιόπιστες και διασταυρωμένες πληροφορίες για τον αριθμό θανάτων, τραυματισμών και συλλήψεων. Επίσης, έχουμε δει, όπως φαντάζομαι και εσείς, βίντεο ελεύθερων σκοπευτών που πυροβολούν διαδηλωτές και έχουμε δει και την επίσημη επιβεβαίωση για τουλάχιστον 7.000 συλλήψεων. Όλα αυτά επισημαίνουν ε, την σοβαρότητα και την κλίμακα των όσων συμβαίνουν. Εμείς δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις. Αντιθέτως έχουμε αντιδράσει και κατηδίαν και δημόσια. Μάλιστα, η πρώτη μου δήλωση ως ύπατος εκπρόσωπος εξ ονόματος των 28 ακόμα κρατών μελών στις 7 Δεκεμβρίου, 9 Δεκεμβρίου αφορούσε ακριβώς τις διαδηλώσεις στο Ιράν. Στη δήλωσή μου αυτή, στη δήλωσή μας αυτή, ξεκαθαρίσαμε ότι παρά τις ε, επανειλημμένες εκκλήσεις ε, για αυτοσυγκράτηση οι Ιρανικές αρχές δυσανάλογα ανταποκρίθηκαν ε, ε, στις διαδηλώσεις και αυτό οδήγησε σε υψηλό αριθμό θανάτων και τραυματισμών. Και πάλι θα ήθελα να τονίσω ότι είτε στο Ιράν είτε οπουδήποτε αλλού η ευρεία χρήση ε, βίας ενάντια σε ειρηνικούς διαδηλωτέ είναι κάτι το μη αποδεκτό. Έχουμε ζητήσει από τις Ιρανικές αρχές και τις έχουμε παρατρύνει να διασφαλίσουν διαφανείς έρευνες ε, που θα διαλευκάνουν τον, τον ακριβή αριθμό θανάτων και τραυματισμών και θέλουμε οι, ε, θύνοντες να λογοδοτήσουν. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζω ότι αυτό το κύμα καταστολής έφτασε ακόμα και στην πρόσβαση στο διαδίκτυο και ότι οι Ρινανοί πολίτες δεν είχαν πρόσβαση ε, στο ίντερνετ, κάτι το οποίο σοβαρά έπληξε την ε, ελευθερία επικοινωνίας. Εμείς θέλουμε να υπάρχει μία ισορροπημένη προσέγγιση και συνεκτική προσέγγιση σε ό,τι φορά το Ιράν για να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα που μας απασχολούν. Φυσικά αυτό συμπεριλαμβάνει και τις ε, μακροχρόνιες μακροχρόνιου προβληματισμού μα ό,τι αφορά την κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επίπεδου μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιράν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με την ε, ε, υιοθέτηση της, της πυρηνικής συμφωνίας από το Ιράν είναι κάτι το οποίο έχουμε θίξει ξανά και ξανά. Επίσης, συστηματικά έχουμε απευθυνθεί στις Ιρανικές Αρχές ζητώντα ε, πρόοδο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την κατάρριξη τη θανατική ποινή, την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των, ε, της πρακτικής των Ιρανών ε, σε ό,τι αφορά την κράτηση των όσων κατέχουν διπλή υπηκότητα. Κάτι το οποίο συνάδει και με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κύριε Πρόεδρε, εξέτοιμα μέλη, κατανοώ πλήρω την σοβαρότητα τη κατάσταση σε ό,τι είχε να κάνει με τι διαδηλώσει και εμεί θα συνεχίσουμε να απευθύνουμε ε, μήνυμα και έκκληση προς τις Ιρανικές αρχές ε, για να αναλάβει συγκεκριμένε ε, ενέργειες στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Ιράν, η οποία δεν αφορά μόνο την Συμφωνία για τα Πυρηνικά. Θεωρούμε ότι οι Ιρανικέ Αρχέ θα πρέπει να σταθούν στο ύψο των διεθνών του δεσμεύσεων και με την ε, διεθνή διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το Διεθνέ Σύμφωνο Πολιτικών ε, και Δημοκρατικών Ελευθεριών. Όπω ε, το δικαίωμα του συνέρχεστε και συνεταιρίζεστε, όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και θέλω να συνεργαστούμε και στο μέλλον για να προαγάγουμε ακριβώς αυτά τα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχουμε αναλύσει διάφορες ε, περιπτώσεις που χρήζουν ε, ισχυρής ε, στάσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Vice President. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μπασέσκου, εκ μέρους του ΕΛΚ, για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει με κάθε τίμημα ε, μια πυρηνική συμφωνία οδήγησε το Ιρανικό καθεστώς να στραφεί κατά του πληθυσμού του και είχαμε ε, τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τη ΣΥΠΑ, όμως ο Αλή Χαμενέη πέρασε στην βίαιη καταστολή των διαδηλωτών σε διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα, σε 31 επαρχίες και σε 130 πόλεις διαδήλωσαν Ιρανοί, όμως ε, πραγματικά ε, το καθεστώς χρησιμοποίησε δυσανάλογη βία εναντίον τους. Σύμφωνα με ε, το Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν, ε, καθεστώς ε, αντιμετώπισε με πρωτοφανή βία τους διαδηλωτές. Ε, περίπου έχουμε 1.500 νεκρούς, από τους οποίους 1.400 είναι επιβεβαιμένοι. Μιλάμε για 10.000 συλλήψεις, 4.000 τραυματίες. Τώρα το καθεστώς ε, αναζητά και συλλαμβάνει ε, όσους συμμετείχαν στις διαδηλώσεις αλλά και τους αρχηγούς επικής αυτοδιοίκησης. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την ε, υποχρέωση να διαμαρτυρηθούμε και να δράσουμε θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στη σχέση της με το Ιράν έχει γίνει δέσμια της πυρηνική Συμφωνίας. Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά και ο λόγος για τον οποίο ε, δεν ε, ε, βλέπουμε ότι το Ιράν, ενώ φιλοδοξεί να γίνει περιφερειακή δύναμη, εμπλέκεται και κόβεται το μικρόφωνο του μιλητή. Συγγνώμη, έκοψα το μικρόφωνο σας, λέει ο Πρόεδρος. Your microphone is cut off. Thank you. Έχω κόψει το μικρόφωνο σας. Our next speaker is Mr. Επόμενος ο κύριος ε, Ντεμπέσα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, με καλώς ήρθατε στο Κοινοβούλιο και σας ευχαριστώ και για το χρόνο που αφιερώσατε σήμερα για να συζητήσουμε όλες αυτές ε, τις περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ, εξ ονόματος Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών, ενστερνίζομαι τη θέση σας και την παρέμβασή σας, η οποία ήταν λεπτομερής και πλήρης. Επίσης, ε, ήταν ιδιαίτερα συνεκτική σε ό,τι αφορά την ε, καταδίκη των γεγονότων ε, στο Ιράν από τον περασμένο Νοέμβρη. Θέλω μόνο να προσθέσω κάποια στοιχεία στο ΣΑΙΠΕ, είπε το εκπρόσωπος. Καταρχήν, επενθυμίσω ότι αυτές οι διαδηλώσει είναι σίγουρα οι μεγαλύτερες που βίωσε ε, το σημερινό καθεστώς ε, στα 40 χρόνια υπαρξής του. Δεν ήταν ειρηνικές οι διαδηλώσεις αυτές, όπως υπόθηκε, ε, και έχουμε κάποιες εκθέσεις από τα Ηνωμένα Έθνη και τη Διεθνή Αμνηστία που μιλούν για τουλάχιστον 300 νεκρούς και 7.000 τραυματίες. Επίσης, ε, πάρα πολλοί έχουν συλληφθεί αυθαίρετα και μπορεί να αντιμετωπίσουν θανατική ποινή. Επίσης, ε, τους αρνούνται βασικά δικαιώματα όπως το να ενημερώσουν ε, την οικογένειά τους και τους αρνούνται και την πρόσβαση σε δικηγόρο. Εγώ πιστεύω ότι το ψήφισμα που θα υιοθετήσει αύριο το Κοινοβούλιο αποτελεί μια απαραίτητη πρωτοβουλία. Ελπίζουμε να συνεισφέρει στο έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή. Η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ακουστεί. Η αντίδραση της κυβέρνησης του Ιράν ήταν πολύ βίαιη και μπορεί να ξεκινήσει τώρα ένας ακόμη πιο καταπιεστικός ή κατασταλτικός κύκλος. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό κράτος και είναι απαραίτητο να έχουμε διάλογο μαζί του. Να, δεν, αμφιβάλλουμε ότι η εξωτερική πολιτική της Ένωση με εσά επικεφαλής θα είναι στο ύψο των περιστάσεων. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Πόριτ για δύο λεπτά εκ μέρους της ομάδας Renew. Ε, μετά από το τελευταίο μας ψήφισμα το Σεπτέμβρη σχετικά με την κράτηση των ε, Ιρανών ε, κατοίκων Ευρωπαϊκή Ένωση Προέλευση, θεώρησα ότι θα έπρεπε να διαμαρτυρηθούμε. Η Ιρανική κυβέρνηση έδειξε μια κατάφορη αγνόηση αυτών των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων. Τον προηγούμενο μήνα είχαμε τις διαμαρτυρίες ε, γιατί έχουν αυξηθεί κατά 50 περίπου τις 100 οι τιμές ε, και αυτή η ειρηνική διαδήλωση ε, λύθηκε με βίαιη καταστολή. Εκατοντάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία τουλάχιστον 304 άνθρωποι, άνθρωποι και παιδιά μεταξύ αυτών δολοφονήθηκαν. Ε, η αρχή και η ελευθερία του συνεταιρίζεστε είναι μια αρχή ε, που δεν γίνεται αποδεκτή. Οι διαδηλωτές στο Ιράν έχουν κάθε λόγο να διαμαρτύρονται, όμως οι Ιρανικές αρχές ε, αντέδρασαν δυσανάλογα και τους προκάλεσαν βλάβες. Είναι λοιπόν καθήκον των κυβερνήσεων να προστατεύουν τους πολίτες και καμία σχέση να έχουν αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Εξάλλου η χώρα έχει αποκλειστεί από online επικοινωνία. Είναι δύσκολο για τους Ιρανούς να διηγηθούν τις ιστορίες τους και αυτό είναι παραβίαση της ε, ελεύθερης ε, έκφρασης. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα όλο και πιο καταπιστικό καθεστώς στο Ιράν. Καταπιέζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι εκτιβιστές ε, γίνονται στόχος γιατί μιλάνε για όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ε, δραστηριοποιηθεί τώρα. Αυτό το ψήφισμα που θα συζητηθεί αύριο απαιτεί να φεθούν αμελητοί ελεύθεροι οι ε, κρατούμενοι και οι ε, εκπρόσωποι της εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνεχίσουν να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ζητήσουν το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να κάνει έρευνα. Τα δικαιώματα των Ιρανών και όλων των υπηκών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πια να περιμένουν. Εκ μέρου των ε, Πρασίνων, αριστερά ο κύριος Ουρτασούν για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάνω από 300 άνθρωποι δολοφονήθηκαν και χιλιάδες ε, κρατήθηκαν ε, στο Ιράν τους τελευταίους μήνες μετά από βίαιη καταστολή από πλευράς Ιρανικών αρχών. Όμως η κυβέρνηση του Ιράν δεν έδωσε καμία πληροφορία για τους κρατούμενους και συνεχίζει να αρνείται όλα αυτά τη βίαιη καταστολή. Ε, η αριθμοί είναι άγνωστοι, δεν γνωρίζουμε και υπάρχουν ισχυρισμοί ότι όσοι βρίσκονται στις φυλακές υπέστησαν κακομεταχείριση. Ανάμεσα στους κρατούμενους είναι φοιτητέ ε, και γι' αυτό το λόγο καλούμε τις αρχές του Ιράν να σταματήσουν αυτή τη βίαιη καταστολή και να διασφαλίσουν ότι θα γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα από τα Ηνωμένα Έθνη για να διευκρινιστούν τα γεγονότα, να διαλευκανθούν και να ε, ζητούν, ζητηθούν ευθύνε από τους ε, υπεύθυνου. Να υπάρξει μια ανεξάρτητη έρευνα για αυτέ τι υπόνοιε για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η οικονομική κατάσταση στο Ιράν επιδεινώνεται λόγω των κυρώσεων και οι τελευταίες διαμαρτυρίες ε, δείχνουν ακριβώς αυτό. Και για το λόγο αυτό επιβραβεύω τις προσπάθειες του ΙΠΑ του εκπροσώπου για να ε, συνεχίσει να ε, χρησιμοποιεί το μόνο εργαλείο που έχουμε για να σταθεροποιήσουμε την περιοχή, το μόνο εργαλείο που έχουμε για να έχουμε διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα. Ως Ευρώπη πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο να διασφαλίσουμε ότι όλοι σέβονται αυτές τις ε, προσπάθειες. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου τώρα της ε, ομάδας ID, κύριε Ρουβιά για δύο λεπτά. Εδώ και δύο χρόνια το πολιτερχικό καθεστώς ε, ε, αμφισβητείται στους δρόμους. Έκλεισαν το ίντερνετ για να παρεμποδίσουν αυτές τις διαδηλώσεις. Το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των προσπαθειών σε σχέση με το Ιράν, την Κίνα και τις ΗΠΑ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα όσα με τη Σαδική Αραβία ε, και τη Συρία. Εμεί καταδικάζουμε ε, την ε, πολιτική του Ισλαμιστικού καθεστώτος και ζητούμε την ελευθερία του ελληνικού λαού. καταδικάζουμε και τις δυτικές δυνάμεις που χρηματοδοτούν τις ε, χώρες που υποθάλπουν την τρομοκρατία. Η δεν είναι μόνο η διπλωματία, γιατί συχνά βλέπουμε ότι οι ελευθερίες αμφισβητούνται και κινδυνεύουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αποτελεσματική, έχει χάσει κάθε αξιοπιστία στην Εγγύη Ανατολή μετά το φιάσκο στη Λιβύη και τη Συρία. Να αφήσουμε ε, τα έθνη της Ευρώπης, που είναι η μοναδική υπέρμαχη ε, των ελευθεριών, να διαλέξουν τη μοίρα τους. On behalf of ECR, ονόματος του ECR, η κυρία Φωτίγκα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Και με τους πλέον συγκρατημένους ε, υπολογισμούς ό,τι αφορά τα θύματα στο Ιράν ε, Πρόκειται για κάτι τόσο ακαριστικό. Χιλιάδες, ε, πάρα πολλοί μάλλον έχουν χάσει τη ζωή τους, χιλιάδες έχουν φυλακιστεί και άλλοι τόσοι έχουν τραυματιστεί. Με βάση αυτή την κατάσταση πρέπει να υψώσουμε τις φωνές μας ε, και είμαι ευγνώμων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί πέρα από τις ε, πολιτικές διαφωνίες είμαστε διατεθειμένοι να ε, ψηφίσουμε ένα κοινό ψήφισμα που θα καταδικάζει το καθεστώς για αυτές τις απώλειες ζώων και να ζητήσουμε από τα Ηνωμένα Έθνη να ερευνήσουν ανεξάρτητα το θέμα. Να ζητήσουμε από το καθεστώς να δημοσιοποιήσει αξιόπιστα στοιχεία ό,τι αφορά τα θύματα, να ε, επιστρέψει τις ορούς των θυμάτων στις οικογένειές τους και να βάλει ένα τέλος στην συνεχιζόμενη ατιμορρησία των υπευθύνων για αυτή την καταστολή. και για τη βία κατά της ε, κοινωνίας στο Ιράν. Ευχαριστώ. Εκ μέρου τη Γκουέ, ε, η κυρία Ένστα ε, για 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Ε, πρώτα απ' όλα, θέλω να ξεκαθαρίσω το εξή, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά. Ανεξάρτητα από το βρίσκεται κανεί ή κάτω από ποιε συνθήκε, δεν μπορεί κανεί να τα διαπραγματευτεί. Παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δολοφονίε ανθρώπων. Για όλα αυτά δεν υπάρχει καμία σχετικοποίηση και δεν μπορεί να υπάρχει σχετικοποιημένη δήλωση. Άρα δηλαδή ε, οφείλουμε να στηρίξουμε τους διαδηλωτέ στο Ιράν, να στηρίξουμε τα αιτήματά τους. Σήμερα δώσαμε το βραβείο Ζαχάροφ ε, και καλό την Ιρανική ε, κυβέρνηση κυβέρνηση επιτέλου να απελευθερώσει τον Νασλουντέ ε, και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είναι ε, απόλυτα ασόβαρο το να ε, λέμε ότι δεν βλάπτει τον Ιρανικό λαό οι αμερικανικέ κυρώσει. Μα βλάπτουν τον λαό και γι' αυτό πρέπει να αρθούν. Οι όξυνση της κρίσης στο Ιράν οφείλεται και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και όποιος ε, παίρνει στα σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να επικρίνει και τις Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίες πρέπει να πάψουν να ασκούν μονόπλευρη πολιτική στη Μέση Ανατολή, γιατί είναι καταστροφική. Όποιος πιστεύει ότι όλο και μεγαλύτερη καταποίηση οδηγεί σε αλλαγή καθεστώτος είναι αφελής. Οι μόνοι που ωφελούνται μέχρι τώρα είναι τα γεράκια του Ιράν. Εκείνοι είναι όμως, ε, αυτοί είναι που παρα παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν. Αλλά αυτοί στηρίζονται. Σας παρακαλώ λοιπόν να τα συνειδητοποιήσετε όλα αυτά. Δεν θα πρέπει να είμαστε μικροπρεπείς, ούτε αφελείς, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ε, στο κατω και γι' αυτό είμαστε εδώ. Εκ μέρου των ε, ε, μη εγγεγραμμένων, ε, ο κύριος Πάτεν για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ ε, για τις εντολοφονίες στο Ιράν και για το ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ε, πολιτικοί κρατούμενοι στο Ιράν ε, που θα πρέπει να φεθούν αμελητοί ελεύθεροι. Αλλά το βασικότερο πρόβλημα στο Ιράν είναι ότι δεν πρέπει το Ιράν να κατασκευάζει πυρηνικά όπλα και να αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή. Τώρα όμως και πάλι έχει αρχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε γρήγορα ε, μια εναλλακτική λύση. Το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών, ε, οι κυρώσει δεν έφεραν τίποτα. Το γεγονό ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει από μόνο του για τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά με τη Ρωσία δεν θα βοηθήσουν. Η εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το θέμα αυτό είναι ένα χάο ε, το Ιράν απειλεί με αντίμετρα κατά ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, βεβαίως και οι μεγάλοι παίκτες δίνουν λίστα προβλήματα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Πολλοί έχουν χάσει το μέτρημα πόσο πολύ προσπαθήσαμε να βρούμε κάποια λύση, αλλά αν θέλουμε το κλειδί στη Μέση Ανατολή είναι να μην υπάρχει υπάρχουν πυρηνικά, να υπάρχει πάλι εμπόριο, να στηριχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ιρανών. Και μόνο οι Αμερικανοί έχουν την δυνατότητα να σκίσουν επιρροή στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ταχύτατα πρέπει να ε, βρει φιλίε στην Ουάσιγκτον, όχι στο Ιράν και νομίζω ότι ε, μπορεί να βοηθήσουν ιδιαίτερα οι σχέσει Μεγάλη Βρετανία με τι ΗΠΑ παρά το Brexit. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ο κατάλογος των ομιλητών εκ μέρου των ε, πολιτικών ομάδων και από τώρα και εξή επιτρέπονται οι μπλε κάρτε. Επόμενο ομιλητής μα, ο κύριο Μάντλ, για 1,5 λεπτό. Αξιότιμε πρόεδρε, αξιότιμε κύριε είπατε εκπρόσωπε, κύριε Μπορέλ, ε, εγώ γεννήθηκα το 79. Και από τότε που γεννήθηκα υπάρχει και το καθεστώς στο Ιράν. Έχουμε την ίδια ηλικία. Παλαιότερα είχαμε μια κατάσταση άσπρο-μαύρο. Σήμερα η κατάσταση ε, προσπαθεί να μην ε, βρίσκεται σε αυτό το ζωφερό τοπίο, αλλά δεν τα καταφέρνει. Και όταν λέμε ότι οι ε, διαδηλώσεις καταστέλλονται με βία, πρέπει να έχουμε κατά νου τις σωστές εικόνες, γιατί το θέμα δεν είναι να τρέχει λίγο αίμα από τις μύτες. Το θέμα είναι ότι έχουμε χιλιάδες νεκρούς ε, που ε, τους έχει ε, νεκροί που οφείλονται στο καθεστώς. Αυτό έγινε πριν από λίγες εβδομάδες. Λίγες εβδομάδες πριν από το 20 του 21ου αιώνα. Τι πρέπει να κάνουμε, να καταστήσουμε σαφές ότι έχουμε μια πυρηνική συμφωνία, όχι γιατί θεωρούμε ότι το καθεστώς είναι αξιόπιστο, ακριβώς γιατί το θεωρούμε αναξιόπιστο. Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε απαρέγκλητα μια συμφωνία για να εμποδίσουμε το Ιράν να καταστήσει κατασκευάσει όπλα πυρηνικής καταστροφής. Γιατί αυτό θα είναι κίνδυνος για ολόκληρο τον κόσμο. Και ω εκ τούτου, κύριε είπατε εκπρόσωπε, σας καλώ ε, να επιβάλλετε σοβαρά διπλωματικές κυρώσεις. Τις ανακοινώσατε εξάλλου στην παρέμβασή σα. Αυτό το χρωστάτε στους Ιρανούς, ε, γιατί πρέπει να αγωνιστούμε και εμείς για τη δική του την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η κυρία Σάντος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αυτό το κοινοβούλιο ξανά τη δραματική κατάσταση στο Ιράν σε λιγότερο από ένα μήνα. Και βλέπουμε επειδή είναι στις τελευταίες εβδομάδες. Η Ιρανική κυβέρνηση όχι μόνο αγνόησε τις εκκλήσεις σε αυτοσυγκράτηση, αλλά ε, κατέστηλε με ακόμη μεγαλύτερη ιδιαιότητα τις ειρηνικές ε, διαδηλώσεις σε όλος της χώρας, ε, που ξέσπασαν λόγω της πολύ σοβαρής οικονομικής και πολιτικής κατάστασης. Έχουμε 304 δολοφονημένους, μεταξύ των οποίων 12 παιδιά σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Έχουμε χιλιάδες συλλήψεις αυθαίρετες ε, και ε, οι κρατούμενοι ε, υφίστανται βασανιστήρια και δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται. Επίση, μπορεί να απεληθούν και με την επιβολή τη θανατική ποινή. Πρόκειται για ρυθμιστικά στοιχεία και γεγονότα τα οποία δεν μπορούμε να τα γνωρούμε. Ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί θεμελιώδε μέρο ε, του διαλόγου που έχουμε με τα άλλα κράτη, αλλά το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και στον πολιτικό διάλογο υψηλού επίπεδου μεταξύ Ιράν και Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιβάλλεται, κύριε Επίτροπε, να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα προκειμένου να πιστούν οι Ιρανικέ αρχέ να αναλάβουν τι ευθύνε του ε, και να σεβαστούν τι ε, διεθνεί συμβάσει που έχουν υπογράψει. Ο κύριος Γκροσέλ για ένα μισή λεπτό. Κυρίες και κύριοι, οι πρόσφατες διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν ε, οδηγήσει σε χιλιάδες φυλακίσεις. Ε, φυσικά μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις για το αν αιτιολογείται η απόσυρση των από την ε, συμφωνία, όμως ε, τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την κτηνοδία και τη βιαιότητα με την, την οποία ασκεί κατά του πληθυσμού. Ε, η Ιρανική κυβέρνηση. Δεν ε, υπάρχει καμία δικαιολογία για τη βία ενός καθεστώτος το οποίο χρησιμοποιεί τις παραστρατιωτικές δυνάμεις και τις κατασταλτικές του δυνάμεις, όχι μόνο στο Ιράν, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από τα πολιτικά και οικονομική της συμφέροντα, πρέπει να, να καταδικάσει τις ε, δράσεις του καθεστώτος δεν θα πρέπει να περικλίνουμε από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κτηνοδία του Ιρανικού καθεστώτος επίσης δείχνει ότι απειλείται ένα θεοκρατικό καθεστώς θα πρέπει να ξέρει ότι αν δημιουργεί, αν χρησιμοποιεί τέτοια καταστολή δεν μπορεί να διασφαλίσει την επιβίωσή του. Μόνο ε, η πολιτική αλλαγή είναι η οδός. Η κυρία Ζερόμ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ποιο λαό θα δεχόταν ε, η τιμή τη βενζίνη να διπλασιαστεί χωρί καμία αντίδραση. Ε, Τι διαδηλώσει του Ιράν κατανοούμε και στη Γαλλία βλέπουμε ε, με τους οδηγούς που αυξάνονται τα διόδια, βενζίνες και ούτω καθεξής, έχουμε τα ίδια. Βλέπουμε ότι είναι απολυταρχικό το καθεστώς, περιμένουμε βελτίωση και πρόοδο σε ό,τι αφορά την, ε, το θεωρητικό χαρακτήρα. Όμως σήμερα τι έχουμε ως μόχλευση. Η, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, και η Γαλλία ε, με δυσαρέσκεια είδαν και την μονομερή απομάκρυνση της αμερικανικής πλευράς από την συμφωνία. Θέλουμε να συνεχίσουμε να σκούμε πιέσει στο Ιράν ε, και να συνεχίσουμε να επιβάλλουμε κυρώσει. Όμως ε, η στρατηγική αυτή δεν είναι αποτελεσματική γιατί είναι πολύ εθνικιστική η κυβέρνηση. Πρέπει να διαμορφώσουμε εκ νέου μια ισορροπημένη σχέση με το Ιράν πριν να αναλάβουμε οποιαδήποτε άλλη ε, πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάιμερς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπατε εκπρόσωπε Μπορέλ. Επιτρέψτε μου να σας μιλήσω για δύο εφήβους. Μίκτα Σφανιάρη, μόλις 14 ετών, όταν την πυροβόλησαν στο κεφάλι οι Ιρανικές αρχές. Η οικογένειά της έψαχνε τρεις μέρες ε, να βρει τη σωρό της. Τα παράλληλα, τα παιδιά όσων ευθύνονται για τον θάνατο της Μίκτα ε, ζουν ανέμελοι στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπου ζουν, ψωνίζουν, ανεβάζουν φωτογραφίες τους στο Instagram ε, και παρακολουθούν ε, στα καλύτερα, μαθήματα στα καλύτερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Χρειαζόμαστε στοχευμένες κυρώσεις κατά του Ιράν, τα μέλη των οικογενειών αυτών των Ιρανικών αρχών πρέπει να γνωρίζουν ότι η πύλη προς την Ευρώπη είναι κλειστή. Να μάθουν οι οικογένειές τους λοιπόν ότι ε, οι οικογένειες των θυμάτων να μάθουν ότι η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό τους. Ευχαριστώ. έχουμε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν ε, θέλω να καταδικάσω την τρομερή καταστολή ε, του καθεστώς των Αγιατολάχ στο Ιράν. Μιλάμε για μια καταστολή που σύμφωνα με αντιφατικά δεδομένα, επειδή το ίδιο το καθεστώς θέλει να αποκρύψει ε, τι κάνει, Μιλάμε για πάνω από χίλιους νεκρούς και πάνω από 7.000 ε, συλληφθέντες και για ε, την δολοφονία 12 παιδιών. Μιλάμε για τρομερή καταστολή και ήθελε το καθεστώς ε, ε, να αποφύγει τις ευθύνες του, μάλιστα κατηγορώντας και τρίτα κράτη. Έκοψε το πρόσβαση διαδίκτυο σε πάνω από 80 εκατομμύρια Ιρανούς και κατηγόρησε τις ΗΠΑ, Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ για την κοινωνική δυσαρέσκεια. Σήμερα από εδώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να πούμε στους Ιρανούς ότι δεν είναι μόνοι δεν είναι μόνοι οι νέοι που διαδηλώνουν στους δρόμους για τις ελευθερίες και τα δικαιώματά τους. Δεν είναι μόνο οι γυναίκες που κάθε Τετάρτη ε, διαμαρτύρονται για την υποχρεωτική χρήση της μαντήλας. Δεν είναι μόνο οι ομοφιλόφιλοι, ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι στη φυλακή. Επίσης ήθελα να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε συνεπείς όταν υπερασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να απευθυνθώ σε κάποια τμήματα της αριστεράς που από ό,τι φαίνεται διαφορετικά ε, υπερασπίζουν τα ανθρώπινα ανθρώπινα δικαιώματα αναλόγως με το που γίνονται αυτές οι υπερβιάσεις. Γι' αυτό θέλω να πω ότι για μένα το αυριανό ψήφισμα μου φαίνεται λυπές και απευθύνω έκκληση να περάσουμε από την απλή καταδίκη στις κυρώσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκούτελαντ, για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν πει ότι τουλάχιστον 7.000 ε, άνθρωποι έχουν ε, συλληφθεί στο Ιράν από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσει τον περασμένο μήνα. Εμείς ζητούμε την ε, άμεση απελευθέρωση αυτών των συλληφθέντων, των συλληφθέντων. Είναι απίστευτο και τρομακτικό να ακούμε για πυροβολισμού διαδηλωτών και φαινόμενα που έχουν χάσει τη ζωή τους τόσοι άνθρωποι και με το κλείσιμο του διαδικτύου ε, αυτό να την κατάσταση παρακολούθησης σε ό,τι αφορά τον ε, αριθμό των ε, θυμάτων και της επιτόπου κατάστασης σε δεκάδες πόλεις. Είναι απαράδεκτο άνθρωποι που απλώς διαδηλώνουν για τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες να ε, δολοφονούνται. Καταδικάζουμε αυτές τις ε, δράσεις και ενέργειες του καθεστώτος. Απαιτούμε να σταματήσει αμέσως αυτή η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ βρίσκεται στο πλευρό του. Θέλω να υπεψηφίσω το ψήφισμα, αλλά πρέπει να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να θίγει το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στι ε, διμερεί και πολυμερεί ανταλλαγές απόψεων. Ευχαριστώ. Η κυρία Ροντρίγε Ράμο. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πατεκπρόσωπε, χωρίς ε, στοιχεία η διεθνή Αμνηστία μιλά για 304 νεκρούς, ε, η Ιρανική Αντιπολίτευση μας λέει για πάνω από 1.000 νεκρούς, 4.000 τραυματίες, 12.000 ε, συλληφθέντες. Και πάλι είχαμε την παρεμπόδιση της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Όμως παρόλα αυτά μας στείλαν κάποιες εικόνες, βίντεο που βλέπουμε να πυροβολούν ε, οι δυνάμεις ασφαλείας ε, από τις εσκεπές, ή από ελικόπτερα κατά των διαδηλωτών. Οι οικογένειες δεν μπορούν να μάθουν ε, συγγνώμη, δεν μπορούν να θάψουν τα παιδιά τους ή τους συγγενείς τους και πριν ε, δύο εβδομάδες βρέθηκαν πολλά πτώματα ε, σε λίμνες και σε ποτάμια. Το Κοινοβούλιο καταδικάζει εκ νέου αυτή την ε, τρομερή καταστολή και ενώνουμε τη φωνή μας με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και ε, ζητάμε μία έρευνα από τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι υπεύθυνοι. Ο απαραίτητος πολιτικός διάλογος με το Ιράν ε, δεν μπορεί να βασιστεί στην ατιμορρησία ε, των δημίων. Ο κύριος Ποσπισίλ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πατεκπρόσωπε. Εγώ είχα καλέσει την κυρία Μογκερίνη στο παρελθόν να υθετήσει μια πολύ πιο αυστηρή στάση απέναντι στο Ιρανικό καθεστώς. Είναι σαφές ότι μια τέτοια χώρα δεν μπορεί να αποτελεί εταίρο μας το καθεστώς ε, δολοφονεί εκατοντάδες ανθρώπους. Θα πρέπει να τα καταδικάσουμε όλα αυτά με απόλυτη σαφήνεια. Ας υιοθετήσουμε μια πιο ριζοσπαστική προσέγγιση απέναντι σε αυτή τη χώρα ε, το Ιρανικό καθεστώς θα πρέπει να ερευνήσει όλα αυτά τα εγκλήματα κατά του ίδιου του, του λαού. Μιλάμε εδώ με μια, για μια πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. Είναι μόνο όμως ένα χαρτί αυτό, εξακολουθεί να ισχύει. Δεν μπορούμε να έχουμε καλές και ορθές σχέσεις με το Ιράν αν συμπεριφέρονται έτσι, πυροβολούν τους ίδιους τους πολίτες τους, οι οποίοι διαμαρτύρονται. Αυτό είναι απαράδεκτο. Κυρία Γκέτα, για ένα λεπτό. Ακούσαμε για χιλιάδες θανάτους που ήδη ήταν κάτι το τρομερό, αλλά έχουμε ακόμα έναν ονομαστικό κατάλογο που είναι ακόμα προσωρινός και μιλάμε για 300 θύματα που έχουν πυροβοληθεί. Αυτό δημιουργεί έναν πανικό, γιατί επίσης αφισβητείται στο εσωτερικό και απορρίπτεται από τα προτεκτοράτα της Λιβύης ε, και του Ιράν. Του Ιρακ. Ε, τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν ε, πέραν των, της ηθικής καταδίκης. Θα πρέπει να προτείνουμε Πρώτα απ' όλα τη διπλωματία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν θα πρέπει να καθυστερήσει πλέον να υποβάλει προτάσει ό,τι αφορά τον προσδιορισμό ζωνών επιρροή, ε, διοργάνωση μια περιφερειακή συνεργασία και θέσπιση εχεγγύων ασφαλεία. Πρέπει να υποβληθούν αυτέ οι προτάσει. Θα χρειαστεί πολλή χρόνο, γι' αυτό και η διπλωματία θα πρέπει να ξεκινήσει ε, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των ομιλητών και τώρα ακολουθεί η διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Βέρ, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, την ε, Δευτέρα Μίλησα και πάλι εδώ σε αυτή την αίθουσα για τον αριθμό των ε, θυμάτων, των θυμάτων που προκάλεσε η βίαιη καταστολή στο Ιράν. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ορισμένα θέματα. Καταρχήν θεωρώ ότι πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξουμε ανεπιφύλακτα την αντιπολίτευση η οποία επιθυμεί την δημοκρατία στο Ιράν. Επίσης είναι απαραίτητο να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με το Ιράν και δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια ε, όπως και οι ΗΠΑ και εμείς θα πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις. Βεβαίως ε, πρέπει να λάβουμε και άλλα συγκεκριμένα μέτρα κατά του καθεστώτος του Ιράν, το οποίο είναι βίο όχι μόνο εναντί των ίδιων πολιτών, αλλά αποτελεί και απειλή στην περιοχή, είναι παράγοντας αστάθειας, ε, αναπτύσσει καινούρια όπλα, όχι μόνο για να απειλεί το Ισραήλ, αλλά και άλλες ε, άλλες χώρες στην περιοχή και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα ήταν λοιπόν λάθος ε, να στείλουμε επιτόπου μία αποστολή στο Ιράν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Δεν είναι στην αίθουσα όμως. Η κυρία Ward. Η Διεθνής Αμνηστία είπε ότι πάνω από 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σκοτώθηκαν και πάρα πολλοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των ειρηνικών ε, διαμαρτυριών στο Ιράν. Το κύμα αυτό διαμαρτυριών είχε σαν αποτέλεσμα επίσης πολλές συλλήψεις 700 φοιτητών, δημοσιογράφων κτλ. Και, τα λοιπά και φαίνεται ότι πέσαν και βασανισμούς. Δεν μπορούμε λοιπόν να καθόμαστε και να μην κάνουμε τίποτα. Είναι σαφές ότι οι Ιρανικές αρχές θέλουν να καταστήλουν κάθε αντιφρονούντα και κάθε αντιπολίτευση. Και όταν μιλάμε για το Ιράν πρέπει να συζητήσουμε επίσης και για τον Τζακαρικλάφτε που επίσης έχει βρεθεί με κατηγορίες και την μέρη που έχει δώσει φοβερές υπηρεσίες έχοντας ε, φροντίσει για τη διάδοση του πολιτισμού του Ιράν. Αλλά εδώ πέρα πρόκειται για ένα διπλωματικό παιχνίδι. Και τέλος θέλω να υπάρξει συνδυτοποίηση για την παρενόχληση δημοσιογράφων και των οικογένειών τους στο Ιράν, ακόμα και αυτών που δουλεύουν για το BBC. Αν είμαστε υπέρ της ελευθερίας πρέπει να την υποστηρίζουμε παντού αυτή την ελευθερία. Η κυρία Ντέιλι, ένα λεπτό παρακαλώ. Η αλληλεγγύη μου εννοείται πηγαίνει πρώτα απ' όλα στα θύματα της καταστολής όπου και αν αυτή λαμβάνει η χώρα, πραγματικά όπου και να λαμβάνει η χώρα και ακούμε για καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν και φυσικά είναι κάτι που καταδικάζω. Το πρόβλημα όμως είναι το εξή. Ακόμα και αν ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, οι καταχρήσει που γίνονται και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μερικές φορές τα υπερβάλλουμε, μερικές φορές όχι. Και ξέρετε τι, πάντα υπάρχουν παραβιάσεις από άλλες χώρες, ποτέ από τις δικές μας από χώρες που έχουν δικιά τους ανεξάρτητη πολιτική, που δεν τους αρέσουν οι Ηνωμένες που έχουν άλλη εξωτερική πολιτική. Φυσικά και πρέπει να στηρίξουμε τα θύματα της καταστολής, αλλά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε μονομερείς όταν πρόκειται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και καταδικάζουμε την καταστολή που γίνεται από τη Ρωσία, την Κίνα ή το Ιράν, αλλά ποτέ από τους φίλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μιλάμε για την καταστολή στους Παλαιστινίους από τους εγκληματίες πολέμου του Ισραήλ. Τότε θα ήμασταν πραγματικοί και σωστοί αν καταγγέλαμε παντού κάθε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ο κ. Καστάλτο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε εκπρόσωποι, συνάδελφοι, τα θύματα που προξένησε η δύναμη ασφαλείας κατά των διαδηλώσεων στο Ιράν ε, είναι περίπου 304 νεκροί, από αυτούς 12 παιδιά και 13 γυναίκες. Αυτοί που έπρεπε να είναι στην πρώτη γραμμή για την να υπερασπίζουν τη χώρα, ε, πυροβολούν το πλήθος, είναι λάθος. Έδωσε την εντολή ο Πρόεδρος και ξεκίνησε μια νέα ε, περίοδο βίας καταστολής. Είχαμε δημοσιογράφους, προσφυγέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φοιτητές, 7.000 που υπήρξαν θύματα. Λοιπόν, δεν μπορεί να μείνει ατιμόρυτο δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε αυτές τις πράξεις που καταδικάζω στεναρά αυτές τις πράξεις. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από την ακριβή βενζίνη που είναι αποτέλεσμα των κυρώσεων των άκρων τιμωρητικών που επιβλήσαν τις ΗΠΑ ε, έναντι ε, του Ιράν και εκείνων που εμπορεύονται με το Ιράν. Αυτό είχε καταστροφικό αποτέλεσμα όσον αφορά τους, ε, το, το πληθυσμό, χωρί να έχει τα αποτελέσματα, τα επιθυμητά, τα πολιτικά. Αυτό είναι κόδων ε, κινδύνου. Εάν πλήττονται τελικά οι πιο αδύναμοι και έχουμε την ελπίδα αυτόν τον τρόπο να επηρεάσουμε αυτού που έχουν την εξουσία. σω αυτό πρέπει να το ξανασκεφτούμε όταν βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα, τα στρεβλά. Εκβάθρων. Ο κύριο Τόμακ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε θα ήθελα να απευθυνθώ προς τον το εκπρόσωπο υπό την ιδιότητά μου σαν μέλος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ευρωκοινοβούλιο. Είπατε εκπρόσωπε, ε, ανήλικοι πέθαναν, νέοι άνθρωποι, δάσκαλοι, ε, μαθητές, φοιτητές. Ήταν όλοι Ιρανοί πολίτες οι οποίοι δεν είχαν άλλο τρόπο να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους παρά μέσω διαμαρτυριών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διπλωματία μας δεν μπορεί πλέον να είναι συνετή και προσεκτική Χρειαζόμαστε αποφασιστική δράση να καταδικάσουμε τα τεκτενόμενα στο Ιράν. Για λόγω της πυρηνικής συμφωνίας δεν μπορούμε να ανεχόμαστε αυτά που συμβαίνουν εκεί. Το Ιράν είναι ένας τόπος αστάθειας και μπορεί να αποσταθεροποιήσει όλη την περιοχή. Συρία, η Εμένη, ε, βλέπουμε τα χέρια του Ιράν παντού και χρειάζεται αποφασιστική δράση. Αυτό ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριο Λόπεθ Ακελάρ, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, δυστυχώς η συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, περισσεύεται πολύ συχνά γύρω από το Ιράν. Η αριθμοί είναι τρομακτικοί. Ε, οι νεκροί είναι πάνω από γύρω στους 300 ε, υπάρχουν πάρα πολλοί κρατούμενοι οι οποίοι φυλακίζονται, βασανίζονται και κινδυνεύουν να θανατωθούν. Όταν ε, μιλάμε για καταστολή ε, των ε, διαδηλώσεων, εννοούμε στην ουσία μια, ένα λουτρό αίματος. Ε, όσον η διπλωματία μπορεί να κάνει πολλά πράγματα όσον αφορά το πολιτικό διάλογο, όχι μόνο με τις αρχές του Ιράν, αλλά και με την αντιπολίτευση του, ώστε να εξασφαλίσει ότι όταν έρθει η στιγμή που να μπορεί να αλλάξει όλη αυτή η πολιτική καταστολή στο Ιράν μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή στο επίπεδο ποιότητας ε, που να υπάρξει μια ελευθερία του, της έκφρασης και ελευθερία της, ε, του θρησκεύματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γουάλλας ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ενώ ε, η, η απάντηση στις ε, διαδηλώσεις δεν μπορεί να ε, δικαιολογηθεί η βία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται κατά των διαδηλωτών και θα πρέπει να την καταδικάσουμε. Επίση, θα πρέπει να καταδικάσουμε τη χρήση βία από, την, από τι ακροδεξιέ κυβερνήσει στη Βολιβία και στη Χιλίου που έχουν θανατωθεί πάρα πολλοί και χιλιάδε έχουν φυλακιστεί. Αυτή η βία η απόκριση ε, είναι ευπρόσδεκτη μόνο από τι ε, ΗΠΑ, οι οποίοι. Ε, όπου ο Μπράιν Χουκ είπε ότι θα πρέπει να θεωρήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα ως σημαντικό θέμα όσον αφορά τη σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν. Γιατί αυτό είναι ένας ε, τρόπος να ασκείται πίεση και να έχουν πλεονεκτήματα όσον αφορά την, ε, τη γεωστρατηγική πολιτική. Η πολιτική κατά του Ιράν οδηγεί τους ε, πολίτες του Ιράν να γίνονται θύματα αυτής της ξένης ε, παρέμβασης. Κύριε Μπορέλ, μπορείτε να αποδεχτείτε κάτι τέτοιο. Η αμερικανική φιλοδοξία είναι να υπονομεύσει τα σχέδια ειρήνευσης στο Ιράν και τον αφοπλισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, χαιρετίζω τους πολίτες της Ευρώπης. Στη συνέχεια έχει το λόγο ο κύριος Μπορέλ. Παρακαλώ. exchange of Αυτή η ανταλλαγή απόψεων ήταν ιδιαίτερα ενημερωτική. Και σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να μάθω περισσότερα για τις απόψεις σας για αυτό το δύσκολο θέμα που είναι οι σχέσεις μας με το Ιράν. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα αγνοήσουμε τους ε, χιλιάδες ανθρώπους που συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες στο Ιράν.